Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να καθίσετε και παρακαλώ και τον κύριο Σμιτ, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Mr. Σμιτ, please, take your seat. Το επόμενο σημείο, παρακαλώ, σας παρακαλώ όσοι κάθεστε όρθιοι είτε να κάτσετε στη θέση σας είτε να βγείτε από την αίθουσα γιατί η συζήτηση συνεχίζεται. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα υλοποίηση και κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Εξ του Συμβουλίου το λόγο έχει ο κύριος Σμιτ. Παρακαλώ κύριε Σμιτ έχετε το λόγο. <laughs> Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, λίγες μέρες πριν τερματιστεί το έτος για την ανάπτυξη